Κίνα και άλλε τέτοιε οικονομίε ε, δεν ασχολούνται καθόλου με το ζήτημα. Και ποιο θα πληρώσει τα σπασμένα με αυτή την ουτοπία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εταιρείε και οι πολίτε. Σα ευχαριστούμε, συνάδελφε Στάσεν. Και τώρα θα περάσουμε στου μεμονωμένου ε, ομιλητές ε, από πλευρά των πολιτικών ομάδων, η κυρία Χάνσλικ.